Προέδρου και η εξέταση των εντολών. Σας ανακοινώνω πως έχουν σχηματιστεί οι εξής κοινοβουλευτικέ ομάδες. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Χριστιανοδημοκράτες, ΕΛΚ, η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κοινοβουλευτική ομάδα της ε, Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ΑΛΔΕ, η ομάδα των Πρασίνων, η Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, Πράσινη, η ευρωπαϊκή Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, η Συνομοσπονδία της ε, Ενωμένης Πράσινης ε, Αριστεράς και Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, GUE-NGL, η ομάδα της Ευρώπης για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 για τον σχηματισμό των ελευθερικών ομάδων έχουν δοθεί